Ε, και η έμπρακτη συμμετοχή στη συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και σας ε, προσκαλώ θερμά να συμμετέχετε και στις συζητήσεις. Θα ήθελα να σας επιθυμίσω ότι για τις ε, διακοινοβουλευτικές επιτροπές η προθεσμία για τις υποψηφιότητες λήγει σήμερα στις 10 το πρωί. Και οι ψηφοφορίες θα γίνουν σήμερα μετά τις 12. Επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα τη Σύνοδο Κορυφής των G20 στο